σε όλο τον κόσμο σε συσχετισμό με τους φόνους των φοιτητών στην Κένια από την τρομοκρατική ομάδα Al-Shabaab. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το λόγο έχει και πάλι ο κύριος Μίμητσα που εκπροσωπεί την κυρία Μογκερίνη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εγώ Συμμερίζομαι τι ανησυχίε σα ε, για του δείχνους συναντήμου των χριστιανών ε, σε όλο τον κόσμο. Ε, είδαμε και τους βορβαδισμούς στο Πακιστάν, τις δολοφονίες στην Ιγυρία, του αποκεφαλισμούς στη Λιβύη, τη συνοχή διωγμών από το ISIS, ανταές στη και στο Ιράκ και την πιο πρόσφατη σφαγή στο Πανεπιστήμιο Γκαρίσα στην Κένια. Όλα αυτά μας δίνουν την εντύπωση μιας πολιορκημένης κοινότητας. Το να στοχεύονται ε, οι χριστιανοί είναι εντελώ απαράδεκτο. Η, ε, βαρβα... βαρβαρική βία και οι απάνθρωπες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται παραδείγματος χάρη από την Λεσεμπέπ, το Άισι, στην Πόκο Χάραμ και οι επιθέσεις ε, κατά του σοβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών και φυσικά ε, κατά της φύσης, ε, της ε, ανθρωπινότητάς μας, ανεξάρτητα από τη θρησκεία μας ή το θρησκευμά μας. Υπάρχουν κτηνοδίες, δολοφονίες, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διενεργούνται από αυτές τις τρομοκρατικές ομάδες κατά των χριστιανών αλλά και κατά άλλων θρησκειών και εθνοτικών ομάδων που δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε στη συζήτηση αυτή. Όπως ε, υπενθυμίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές για την ελευθερία της θρησκευτικής πεποίθησης, η θρησκεία τον Ιούνιο του 2013, όλα τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες, σε θρησκευτικές κοινότητες, θα πρέπει να μπορούν να λατρεύουν ελεύθερα και να ασκούν τη θρησκεία τους ελεύθερα, ατομικά ή σε κοινότητα μαζί με άλλους, ε, χωρίς να υπάρχει μισολοδοξία και επιθέσεις. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να παραβιαστούν αυτές οι αξίες, να τεθούν σε κίνδυνο. Αυτό ισχύει για ανθρώπους όλων των θρησκευμάτων, ήταν ενό θρησκεύματος και φυσικά αυτό ισχύει και για τους χριστιανούς. Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχάσουμε ότι το πρώτο θύμα της τρομοκρατίας είναι οι μουσουλμάνοι Στις ε, αραβικές χώρες. Ε, θα πρέπει να μην πέσουμε ε, στην λογική μιας, μιας σύγκρουσης πολιτισμών. Ο βασιλιάς Ιορδανίας μας τα υπενθύμησε όλα αυτά όταν απευθύνεται την ομιλία του σε αυτόν τον ε, οίκο. Είπε ότι οι επιθέσεις ε, κατά των χριστιανών και κατά μειονοτήτων σε ορισμένε χώρες είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας ε, όπως και κατά του Ισλάμ. Οι Άραβες χριστιανοί αποτελούν σημαντικό τμήμα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντός μας, είπε ο Βασιλιάς. Σήμερα στο νότιο τμήμα της Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια σειρά κρίσεων και σειράξεων που υπάρχει δυνατότητα να διαχειθούν. Είναι σημαντική η συνεργασία μας με τους Άραβες εταίρους μας αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις απειλές που βιώνουμε σήμερα. Απειλέ στην ασφάλεια φυσικά συμπεριλαμβάνουν και την τρομοκρατία των τζιχαντιστών και το, διεθνές, το διεθνικό έγκλημα. Πρέπει να συνεργαστούμε και για την προστασία των μειονοτήτων και που ε, προκαλούν και για τις αιτίε που προκαλούν αυτές τις κρίσεις συμπεριλαμβανομένους και της λήψη υποψής της κατάστασης ε, των νέων γενεών. τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου για την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας ε, θέτουν με ακρίβεια μία σειρά δράσεων για να καταπολεμήσουμε ε, το ριζοσπαστισμό και την τρομοκρατία. Εδώ έχουμε σχέσεις, διμερή συνεργασία, πολυμερή συνεργασία ε, σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις κυβερνήσεις αλλά και με ε, τις τοπικές κοινότητες, υποστηρίζοντας και το διάλογο μεταξύ των θρησκευμάτων. Αλλά θα ήθελα να επανέλθω στην τελευταία επίθεση στην Κένια. Αυτή η κτηνόδες επίθεση είναι η τελευταία και η πιο θανατηφόρος από τις επιθέσεις που έγιναν στην Αλσεμπά από την Αλ Σαμπάμπ στην Κένια τους τελευταίους 18 μήνες. Τρομοκρατικές δράσεις ε, έχουν ε, δυστυχώς Γίνει κάτι συχνό στην Κένια και βλέπουμε μια πυλή να αυξάνεται στο κέρας της ε, Αφρικής. επίθεση στην Καρίσα ε, ήταν ε, πιο σκληρή και ίσως υπήρχε έμπνευση από τις μεθόδους της Μπόκο Χάραμ ή του Ισλαμικού κράτους. Η στόχευση συγκεκριμένη των χριστιανών είχε γίνει και σε προηγούμενες επιθέσεις αυτή η λεγόμενη τάση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική παρά το γεγονός ότι εκπρόσωποι από τη μουσουλμανική κοινότητα της Κένιας τοποθετήθηκαν κάθετα και καταδίκασαν την επίθεση υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να υπάρξει περαιτέρω ανταγωνισμός και διαίρεση μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων και φυσικά αυτό είναι ο στόχος των δραστών. Γι' αυτό είπα ότι εκπρόσωπος Μογκερίνη αναφέρθηκε στις δηλώσεις της 3 ε, Απριλίου στο εξή. Όταν γίνεται επίθεση στους φοιτητέ στον Καρίζα με το θάνατο 147 νέων ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών άλλων τρομοκράτε, έδειξαν ότι είναι αποφασισμένοι να υποσκάψουν ε, την εκπαίδευση, να προκαλέσουν σύγκρουση μεταξύ θρησκευτικών ε, ε, πεπιθήσεων και να απειλήσουν την σταθερότητα και την αξιοπρέπεια τη χώρα για όλου του πολίτε. Έχουμε ένα παγκόσμιο πρόβλημα με τη ριζοσπαστική και τον εξτρομισμό και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την απομόνωση και ενώ χρειάζεται παγκόσμια προσέγγιση θα πρέπει οι λύσεις να αφορούν την κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά. Πέρα από το να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σε εθνικό επίπεδο, το να επανεφεύρουμε παγκόσμιες στρατηγικές, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να χαρτογραφήσει και να κατανοήσει καλύτερα πώς η ριζοσπαστικοποίηση λειτουργεί μεμονωμένα σε διάφορες χώρες όπως την Κένια και σε κοινότητες. Αυτό προκειμένου να βαλτιώσουμε την απάντησή μας και να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ακολουθούν οι ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων και οι ομιλήτες. Ενάμιση λεπτό από το ΕΛΚ είναι η κυρία Τερέσα Χιμένεθ Βεσέριλ Μπάριο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε την περασμένη Μεγάλη Πέμπτη πολλοί από εμά είχαμε πάει στην εκκλησία ελεύθερα. Εκείνη τη στιγμή ακριβώς ένα πανεπιστήμιο στην Κένια, η τρομοκρατική ομάδα Al-Shabaab επέλεγε χριστιανούς φοιτητές για να τους δολοφονήσει. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό τι ανίποτη φρίκη αισθάνθηκαν αυτοί οι νέοι όταν τους ξεχώρισαν από τους ε, συμφοιτητές τους ε, για να τους σκοτώσουν, για να πεθάνουν επειδή ήταν χριστιανοί. Τι αγωνία ε, αισθάνονται οι γονεί των κοριτσιών που απήχθησαν στην Ιγυρία σε ένα χριστιανικό σχολείο ή η απόγνωση ε, των χριστιανών τη Μέση Ανατολή που πρέπει να φύγουν από τα σπίτια τους και να τα εγκαταλείψουν αν δεν θέλουν να πεθάνουν. Γι' αυτό το Λαϊκό Κόμμα έβγαλε ένα ψήφισμα όπου ε, καταφέραμε να συμπεριλάβουμε μαζί με αυτέ τι φρικαλαιότητε στην Κένια ε, τον αριθμό και τους, το, όνομα και τους διωγμούς των χριστιανών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ήθελαν οι άλλες πολιτικές ομάδες ούτε καν να διαπραγματευτούν μαζί μας. Ε, ήθελα να βγάλουμε ό,τι έκανε αναφορά σε χριστιανούς, σε ονόματα. Εγώ αρνήθηκα και κάναν άλλο ψήφισμα οι άλλοι. Από 39 παραγράφους ε, γίνεται λόγος για τους χριστιανούς μόνο σε δύο, ενώ στο δικό μας ψήφισμα γίνεται λόγος για όλες τις διώξεις, τους διωγμούς και τις παρενοχλήσεις που υφίστανται ανά τον κόσμο οι χριστιανοί. Αξίζει ε, ε, στο μέλλον ε, να στραφούμε λένε οι άλλες ομάδες. Όχι κύριοι, κάθε ώρα ε, που περνάει χάνει ένας χριστιανός τη ζωή του. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν είναι συμπλεγματικό, δεν κάνει διάκριση ανάμεσα σε ε, πρώτης και δεύτερης κατηγορίας θύματα. Να υποστηρίξετε το δικό μας ψήφισμα γιατί εμείς υποστηρίζουμε όλους τους χριστιανούς που διώκονται αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια από τους σοσιαλδημοκράτες και πάλι για 1,5 λεπτό είναι η κυρία Ελένα Βαλενθιάνο καταδικάζουμε οποιαδήποτε βία και διάκριση που βασίζεται στη θρησκεία. Οποιαδήποτε θρησκεία. Το καλύτερο αντίδοτο στον εξτρεμισμό είναι η παιδεία και η εκπαίδευση και γι' αυτό το Al-Shabaab χτύπησε πανεπιστήμιο. Και είναι γεγονός ότι έλεγε κάποτε ε, ένας πανεπιστημιακός που σώθηκε είπε ότι αυτό δεν θα ακουστεί πουθενά στον κόσμο γιατί δεν σκότωσαν κανένα λευκό. Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης είναι γεγονό ότι το είδαν πολύ περιθωριακά αυτό το θέμα της φαγής στην Κένια. Και γι' αυτό χρειάστηκε να λανσάρουν οι ίδιοι φοιτητέ ε, μία εκστρατεία, ότι 147 δεν είναι απλώς ένα νούμερο και, είπαν και ανέφεραν και τα ονόματα όλων των νεκρών. Εμείς παραγνωρίζουμε και αγνοούμε την κατάσταση σφόδρα στη χώρα αυτή Ήδη με την ανεξαρτησία της Κένιας υπήρχε μεγάλη σύγκρουση βορρά και ε, νότου ε, ε, με τι υπόλοιπε περιφέρειες και την πρωτεύουσα. Ε, το Ναϊρόμπι και η Γκαρίσα ήταν πολύ μακριά και η Σομαλία ήρθε να επιδεινώσει τα πράγματα. Τώρα οι τρομοκράτε του Αλ Σαμπάπ ε, δηλώνουν ότι είναι ένα πόλεμο αυτό κατά τη Κένια και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει ακριβώ την Κένια για την ασφάλειά τη, για να ελέγξει τα συστήματα και τα προβλήματα ασφαλεία που αντιμετωπίζει. Να του βοηθήσουμε να δουν και τις σχέσεις του με τη Σομαλία. Εμείς λέμε να τους δώσουμε και πολιτική στήριξη, αποφασιστική και μέσα και πόρους. Γιατί είναι ένας πόλεμος που έχει κηρυχθεί απέναντι κατά της Κένιας και κατά όλων μας σε τελική ανάλυση. Ευχαριστώ πολύ από τους φιλελευθέρους για ένα λεπτό τώρα ο κύριος Άντζελ Τζαμπάνσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, τη συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Αναμφίβολα γίνηκαμε μάρτυρες ενός τραγικού περιστατικού, δηλαδή μιας δολοφονίας εξαιτίας της θρησκείας, εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν χριστιανοί. Δεν είναι δύσκολο να το αντιληφθεί κανείς αυτό, ότι ο στόχος των διαγμών ήταν οι χριστιανοί. Και ο λόγος που συνέβη αυτό είναι η επέμβαση, η σχέση, εν πάση της Κένιας με τη Σομαλία. Ο Ισλαμικός φονταμενταλισμός ενισχύεται σε κράτη του, της περιοχής του κέρατος της Αφρικής και θα πρέπει ενωμένοι να τον καταπολεμήσουμε με βάση τις ε, ευρωπαϊκές αρχές, αυτές που βρίσκονται στο στόχο είναι οι αξίες της Ευρώπης και ο τρόπος ζωής μας. Αυτό έγινε νομίζω πολύ ξεκάθαρο πια. Δεν αρκούν τα ψηφίσματα, θα έπρεπε να αναλυφθεί στρατιωτική δράση στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Για δύο λεπτά από τους φιλελευθέρους, ο Ρίκε Καλβέτη Σαμπών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φυσικά ε, ε, ε, Είμαι πολύ ευαίσθητος απέναντι στο θέμα του διαγμών των χριστιανών σε όλο τον κόσμο και φυσικά θα βοηθήσω όλους όσους προωθούν ένα ψήφισμα. Αλλά αυτού όμως η πρόθεσή μας ως ομάδα των φιλελευθερών είναι να επικεντρωθούμε στην δολοφονία των φοιτητών στην Κένια, στον Καρίσα, μια δολοφονία που βασίστηκε φυσικά ε, σε λόγους θρησκευτικού, αλλά και σε εθνοτικούς λόγους και φυσικά και λόγω του πολύ παλαιού πολέμου που υπάρχει ε, στην περιοχή αυτή του κόσμου μεταξύ όσους ε, κατοικούν στην Σομαλία απέναντι στους γείτονές τους και πολύ περισσότερο κατά των δυτικών αξιών, κατά μια σειρά δυτικοποιημένων φοιτητών και τελικά κατά των δημοκρατικών αξιών. Και εμείς θα θέλαμε ε, το ψήφισμα μας ε, να δώσει έμφαση σε αυτή τη συγκεκριμένη τρομερή πράξη για να πούμε ότι η Ευρώπη ε, δεν μπορεί ε, να δέχεται κάτι τέτοιο όπως κάνει το ίδιο και στο Μάλι και αλλού. Θα πρέπει να προστατεύουμε οποιαδήποτε μειονότητα από τους διωγμούς και θα πρέπει να εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό. Θα πρέπει να εμπλακεί επιτόπου με εκπαιδευτές, ε, με ανθρώπους οι οποίοι θα είναι ειδικοί και που με τη βοήθεια των αφρικανικών στρατευμάτων θα προσφέρουν βοήθεια αλλά και θα εμποδίζουν τέτοιου είδους δολοφονίες και διωγμούς που στρέφονται κατά των αξιών που υπερασπιζόμαστε. Αυτό το σκοπό επιδιώκουμε με το ψήφισμα και αύριο θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια για ένα λεπτό από την ελωτική Αριστερά, η Λίντια Σένα Ροντρίγκε. Ευχαριστώ. Καταρχήν, θα ήθελα να σας πω ότι καταδικάζουμε πλήρως ε, τις ε, δολοφονίες και τις επιθέσεις της Αλσαμπάκ στο Πανεπιστήμιο της Γκαρίς. Επίσης να εκφράσουμε την πάσα αλληλεγγύη μας με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δράσει με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να καταπολεμήσει τις βαθιές ρίζες των σειράξεων και που δημιουργούν καταστάσεις που ευνοούν ε, τη δημιουργία ομάδων όπως η Αλσαμπάκ. Πιστεύουμε ότι αν δεν είναι κατάλληλη απάντηση να επικεντρωθούμε στα στρατιωτικά μέσα. Ε, η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σομαλία το 1992 με τρομερές συνέπειες που ακόμη πληρώνουν οι λαοί της περιοχής σήμερα ευθύνη των παλαιών απικιακών δυνάμεων στη λαϊλάτηση των φυσικών πόρων του κέρατος της Αφρικής και στην αρπαγή των δεών, η φτώχεια. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι οι περισσότεροι, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στην Κένια ζει κάτω από το όριο τη φτώχεια, χιλιάδες πρόσφυγες στην εσημότητα των παιδιών, πείνα, και δεν περνά η λύση από στρατιωτικέ επιχειρήσει ούτε του ΙΕ ούτε, ούτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη, ούτε των ΗΠΑ. Θα πρέπει να σταματήσει η λελάτιση τη Αφρική. Θα πρέπει να ολοκληρώσετε και θα πρέπει να σεβαστούν την κυριαρχία των λαών έτσι ώστε αυτή να είναι η κυρίαρχη των πόρων του αλλά και τη μοίρα του. Σα ευχαριστώ. Um, Κοιτάξτε, θα σας παρακαλούσα να τηρείτε το χρόνο σας και να μην μιλάτε και τόσο γρήγορα για να σας προλαβαίνουν οι διερμηνείς. Όταν μιλάτε με τέτοια ταχύτητα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο. Παρακαλώ, αν θέλουν να σας καταλάβουν οι συνάδελφοί σας. Η κυρία Χόιμπουχ για 1,5 λεπτό εξ ονόματος των Φρασίν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι επιθέσεις δολοφονικές στην Κένια θα πρέπει να καταδικαστούν σφοδρότατα. Πάντα ε, ορισμένες ομάδες θέλουν να αυξήσουν τη δύναμή τους εις βάρος κάποιων άλλων. Η Al-Shabaab είναι Ισλαμική πολιτοφυλακή και δεν διστάζει να χρησιμοποιεί τέτοια μέσα και θρησκευτικά για να προσπαθήσει να αποσταθεροποιήσει τη Βόρεια Κένια. Γνωρίζουμε ότι η ομάδα Al-Shabaab έχει κάνει συνειδητά ε, αυτές τις επιθέσεις σε χριστιανούς της Κένιας για τους ανωτερολόγους αλλά ξέρουμε ότι και στην ίδια τη Σομαλία δεν διστάζουν να επιτίθεται και να σκοτώνουν γυναίκες, παιδιά, μαθητές, φοιτητές και μουσουλμάνους. Εδώ χειραγωγείται και χρησιμοποιείται η θρησκεία και δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση. Στο ψήφισμά μας θέλουμε να εστιάσουμε στην Γένεια βασικά και ε, για να το κάνουμε και θα πρέπει να θυμηθούμε την κατάσταση που επικρατεί στην Κένια, ιδιαίτερα στη Βόρεια Κένια, είναι άκρος ασταθής και οι ε, αρχές ε, της χώρας δεν συμπάσχουν πάντα με τις Ισλαμικές μειονότητες και τις προστατεύουν. Ε, αυτό υποδαβλίζει και κριτική και μίση και πάθη και προσπαθεί να κερδίσει δύναμη Αλ Σαμπάμπ. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει απολύτως και πηγόντως να το αποτρέψουμε. Ευχαριστώ συνάδελφοι για ένα λεπτό από την ομάδα του, ο κύριος Καστάλτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ε, είδαμε ότι δολοφονήθηκε εκεί το μέλλον της χώρας με τη δολοφονία σχεδόν 150 φοιτητών όμως ε, δεν ε, είδαμε τους ηγέτες να κάνουν κάτι, να βγαίνουν στο δρόμο μάλλον για το θέμα του Σερλί κάποιοι είναι περισσότερο ή λιγότερο Σερλί βλέπουμε ότι το θέμα αυτό γεννήθηκε από την μαζική μετανάστευση από τις Σομαλία. Ε, είχαμε 150.000 Σομαλούς ε, θύματα. Ε, η τρομοκρατία εποφελείται αν δεν μπορέσουμε να παρέμβουμε για να εξαλείψουμε τη φτώχεια τότε δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη τρομοκρατία. Είναι η πρώτη σύμμαχο της τρομοκρατία η φτώχεια, όπω βλέπουμε και με το παράδειγμα της συγκρούση των πολιτισμών και ακούσαμε ότι το επιθύμησε και ο Πάπας η φτώχεια ε, είναι ο πρώτη σύμμαχος ε, της τρομοκρατίας ενώ η αξιοπρέπεια είναι ο χειρότερος εχθρός. Για... Ευχαριστούμε για ένα λεπτό η Μάρα Μπιτσότου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η το, η των χριστιανών φοιτητών στην Κένια είναι ε, μια τραγωδία. Οι φοιτητέ αυτοί, λόγω απλώ τη θρησκείας του, ε, είναι ένα μικρό μέρο μόνο αυτών που έχουν χάσει τη ζωή του για ένα θέμα που, κάνουν, ε, που η Ευρώπη κάνει όταν το βλέπει. Είναι ε, άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή του με σταύρωση, με εκτέλεση, με φρικτού τρόπου, χιλιάδε ανά τον κόσμο και ε, φαίνεται ότι ακόμα και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι συνένοχοι αφού αδιαφορούν. Μιλάμε για μια γενοκτονία, για την άνεξη θρησκεία του ριζοσπαστικού Ισλάμ που διακηρύσει το μίσος. Εμείς οι χριστιανοί για αυτούς τους αδερφούς μας χριστιανούς δεν έχουμε ούτε δικαίωμα να ζούμε. Θα έπρεπε να σβηστούμε και να, εφόσον δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνε μας. Η Ευρώπη λοιπόν υποτιμά την κατάσταση αυτή. Γιατί η Ευρώπη δεν υπερασπίζεται τις δικές της χριστιανικές ρίζες, την ιστορία της. Γιατί δεν δρά, γιατί δεν αντιδρά, γιατί δεν κάνει τίποτε για να πάψει αυτή την εξόντωση. Ε, σας απευθύνω λοιπόν έκκληση, μία οικησία συνάδελφοι. Μην αφήσουμε το αίμα των αθώων να χύνεται στο όνομα του Αλάχ. Ευχαριστούμε ο κύριος Χέλβενη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ Ε, καλή ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό, διότι εδώ χάσαν τη ζωή τους ε, ένα σωρό φοιτητές για να ευαισθητοποιηθούμε στο Πανεπιστήμιο αυτό της Κένιας. Μιλάμε για απολύτως αθώους ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν θύματα των ε, τρομοκρατών της Αλσαμπάπ. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ε, τι μπορούμε να κάνουμε για όσους μειώνουν τη σημασία αυτού του γεγονότος σε πρώτη φάση. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν διωχθεί, έχουν θανατωθεί. Μιλάμε για μειονότητες οι οποίες ε, διώκονται και η Ευρωπαϊκή Ένωση απλώς κοιτάζει αδιάφορα. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με μια ενιαία φωνή για το θέμα αυτό και να υψώσουμε την φωνή αυτή κατά τέτοιων ε, αιματηρών επεισοδίων. Θα πρέπει να το δούμε όχι ως θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή θρησκείας απλώς, αλλά ένα θέμα σεβασμού του ανθρώπου, της ανθρώπινης ζωής. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας μπροστά σε όσα συμβαίνουν. Πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε οι άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους και να διώκονται για λόγους ε, θρησκείας, θρησκευτικούς. Θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη και αυτό πιο συγκεκριμένα αφορά την δίωξη χριστιανών. Είναι σαφές ότι πρέπει να αντισταθούμε σε κάθε είδους τρομοκρατική ενέργεια. Ζούμε σε ένα κόσμο λαϊκής πίστης, κοσμικό και θα πρέπει οι αξίες αυτές να είναι αξίες που θα προσπιστούμε. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό κυρία Κέντερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Άμος, Θέι, Ελίζαμπεθ, Έντουαρτ, περίπου 150 ονόματα. Άνθρωποι, φοιτητές, νέοι, ελπίδες που χάθηκαν δεν είναι απλώς ε, αριθμοί που καταγράφονται σε ένα μακρύτερο κατάλογο. Σήμερα αποτείμε τιμή στα θύματα που αντιμετώπισαν με ε, τόλμη τον ε, Ισλαμικό ριζοσπαστισμό που ξαπλώνεται σε όλη την Αφρικανική Ήπειρο. Η τρομοκρατία εξ ονόματος της Άλλη shabaab στο κέρα της Αφρικής σημαίνει την απώλεια της νεολαίας. Μια νεολαία που όμως ατενίζει το μέλλον και θέλει την εκπαίδευση για τις μελλοντικέ γενιές. Σήμερα ζητούμε παρέμβαση με πυγμή για να αντιμετωπίσουμε την τυφλή βία, την εξετρεμιστική βία, διότι με τα εκατοντάδες θύματα καθημερινά στον αγώνα αυτό, τελικά διακυβεύεται το μέλλον μιας ολόκληρης υπήρου. Θα πρέπει να δούμε τα βαθύτερα αίτια του κακού, που έχουν να κάνουν με τη ριζοσπαστικοποίηση. Γιατί ο ακραίος Ισλαμισμός ε, συνάδει με την περιθωριοποίηση, τη φτώχεια, γιατί δεν αντιμετωπίζουμε τη διακριτική μεταχείριση κατά των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων εντός μιας χώρας. Ε, ε, πάλι κατά της τρομοκρατία δεν μπορεί να αφορά μόνο την γένεια όμω. ή να είναι ένα πρόσχημα για να καταπιεστούν οι ελευθερίε των πολιτών. Κάθε οπισθοχώρηση ω προ τον εκδημοκρατισμό μια χώρα είναι μια νίκη που κερδίζει η τρομοκρατία. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τι προκλήσει, τι κοινέ αξίε τη ε, σύγχρονη κοινωνία που βασίζονται στι θεμελιώδει αξίε, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Άμο, Φέιθ, Ελίζαμπεθ και Έντουαρτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Υπενθυμίζω και πάλι σε όλους τους συναδέλφους παρακαλώ να μιλούν με μια ταχύτητα που να επιτρέπει και στους διερμηνείς να μεταφράζουν για να καταλαβαίνουμε τι λέτε. Ένα λεπτό, Ρούζα Τόμασιτς. Ευχαριστώ πολύ μου. Πρέπει να θυμηθούμε και να καταλάβουμε όλοι ότι η τρομοκρατία δεν δικαιολογείται από αδικίες που μπορεί να έχουν γίνει έναντι χωρών, έναντι μιας εθνοτικής ή θρησκευτικής ομάδας. Όλοι αυτοί που δικαιολογούν με αυτόν τον τρόπο τη βία την οποία διαπράττουν πρέπει να θέσουν το ερώτημα. Τι έφταιγαν αυτοί οι 147 νέοι που δολοφονήθηκαν. Ήταν μήπως απεικιοκράτες, ποιον είχαν σκοτώσει. Ήταν νέοι οι οποίοι ήθελαν απλώς να σπουδάσουν και ήθελαν να μπορέσουν να ζήσουν. Το μόνο του σφάλμα είναι ότι ήσαν χριστιανοί. Χριστιανοί λοιπόν, που γι' αυτό το λόγο σε όλο και περισσότερα μέρη του κόσμου δεν μπορούν να ζουν. Εκεί που υπάρχει αυτή η τρομοκρατία. Σε πολλά μέρη του κόσμου οι χριστιανοί φεύγουν. Πρέπει να θυμηθούμε ποιες είναι οι αξίες μας. Οι αξίες μας ε, πρώτα απ' όλα είναι χριστιανικές αξίες. Και πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτό που χρειάζεται, ώστε αυτές οι αξίες να μπορέσουν να συνεχίσουν εκεί που είναι εδώ και 2.000 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ δύσκολο να βρω λόγια για αυτά τα τραγικά γεγονότα. Πολλά υπόθηκαν και τα συνυπογράφω. Επίτροπε, αναφερόμενο στην ομιλία σα πρέπει να πω ότι συμφωνώ με όλα όσα είπατε για τι διώξει των χριστιανών και για την Κένια. Αλλά Υπάρχει κάτι όμως που θα προτιμούσα να υπήρχε στην ομιλία σας. Μου έλειψε. Αν μπορείτε να μιλήσετε γι' αυτό. Μιλήσατε για, τις, για τα πορίσματα του Συμβουλίου για τρομοκρατία, για συγκεκριμένες περιπτώσεις και συγκεκριμένες λύσεις. Αλλά σταματήσατε λίγο πριν από το να μας εξηγήσετε ποια είναι η αντίληψή σας για τα ποια διδάγματα έχουμε εξαγάγει. Τι έχει γίνει έκτοτε. Τι έκαναν οι υπηρεσίες σε σχέση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Κένιας. Τι μπορούμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε θεσμούς. Τι χρειάζεται. Ποια συγκεκριμένα βήματα μπορείτε να αναλάβετε για να αποφύγουμε την γεγονότα στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής, ένα λεπτό. Η Νες Χριστίνα Ζούμπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ισλαμιστική βία των ομάδων όπως όλοι στην Κένια είναι απαράδεκτη θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει στρατηγική ε, κατά της θερμοκρατίας, αλλά όχι βάσει ρατσιστικών και ξενοφοβικών αντιλήψεων. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναλάβει τη μερική ευθύνη που αναλογεί στο φαινόμενο αυτό. Είναι πολλά τα αίτια που προκαλούν τέτοιες καταστάσεις, τη ροζοσπαστικοποίηση και στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και στο κέρα της Αφρικής. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε με ενισχυμένες λύσεις ε, τα φαινόμενα αυτά όπως με πρωτοβουλίες σαν αυτή που πρώτα είναι η ομάδα μα. Στην Κένια και σε άλλε αφρικανικέ χώρε θα πρέπει να βασιστούμε σε αρχέ μη παρέμβαση στην ε, σεβασμό τη κυριαρχία, τη ελληνική κυριαρχία των χωρών και να ανταλλάξουμε τα όσα δίνουμε στα πλαίσια των συμφωνίων ελεύθερου εμπορίου με άλλε στρατηγικέ. Λόγου χάρη την ενίσχυση τη αναπτυξιακή συνεργασία με τι χώρε αυτέ τη Αφρική. Θα πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη και στήριξη τη εκπαίδευση, τη υγεία και τη οικονομία. Δηλαδή να λυθούν τα κοινωνικά προβλήματα που ταλανίζουν τι χώρε αυτέ και είναι οι ρίζε του προβλήματο. Ευχαριστώ πολύ. Ενάμιση λεπτό, Τζόναθαν Σίγουρα όλοι εδώ αισθάνονται οργή και θλίψη για τις πρόσφατες δολοφονίες αυτών των χριστιανών φοιτητών σε Πανεπιστήμιο της Κένια. Οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε αυτή η επίθεση είναι εξαιρετικά τρομακτικές. Δεν μιλάμε για τυχαία βία. Αντίθετα, τους χριστιανούς αυτούς φοιτητές τους χώρισαν τους υπόλοιπους και τους δολοφόνησαν. Και θυμάμαι τι είπε ο Απόστολος Παύλος προς Τιμόθεο. Όσοι θέλουν να ακολουθήσουν ε, μια χριστιανική ζωή στα πλαίσια των διδαγμάτων του Ιησού θα διωχθούν. Νομίζω ότι με το δυτικό τρόπο σκέψης είναι εύκολο κανείς να ξεχάσει τις, τις τρομακτικές διώξεις που αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο σε σχεδόν καθημερινό επίπεδο τουλάχιστον σύμφωνα με τη φιλοθροπική οργάνωση Open Doors. Οι επιθέσεις αυτές στην Κένια μπορεί πραγματικά να μας κατατρώμαξαν, αλλά δεν αποτελούν ε, μοναδικό φαινόμενο. 28 χριστιανοί ε, βρίσκονταν ε, στην Κένια, στο Μαντάρι, σε ένα λεωφορείο το οποίο πήχθη, τους κατέβασαν το λεωφορείο και τους δολοφόνησαν. Το ίδιο συνέβη και άλλη μια φορά. Ένας καθολικός παπάς τον Ιανουάριο την ώρα που έφυγε από τη λειτουργία αποκεφαλίστηκε. Και μην ξεχνάτε τι έγινε και με την επίθεση στο εμπορικό κέντρο στο Ναϊρόμπι. Ναι, είπαμε, ε, εξοργιστήκαμε από τη δολοφονία στην εφημερίδα Charlie Hebdo. Όταν όμως έχουμε τέτοιες επιθέσεις στην Αφρική, ξέρετε πως είναι εξίσου τραγικές με αυτές οι οποίες λαμβάνουν χώρο πιο κοντά σε εμάς. Γεωγραφικά για ένα λεπτό θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σαν Φράουζερ. Oui, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη μαρτυρία τους όπου βλέπετε ομόφωνα όλοι οι παρεμέροντες να συμφωνούν η φρικτή δολοφονία στην Καρίσια των 148 φοιτητών πέραν της καταδίκης πρέπει να μας ε, φέρει αντιμέτωπος με την αλήθεια. 150 έως 200 εκατομμύρια χριστιανοί θανατώνονται ανά τον κόσμο λόγω της πίστης τους. Είναι η δεύτερη από, τους πρώτους, ε, από τις δύο κοινότητες που βασανίζονται για τη θρησκευτική τους πίστη, για τη θρησκευτική τους πίστη τις πεπιθήσεις τους. Ε, δεν αποσιωπάται βεβαίως το στοιχείο αυτό, αλλά υπάρχουν εφημερίδες που αρνούνται τη σφαγή αυτή και το ερώτημα είναι εάν θα πρέπει να ε, αδιαφορήσουμε για αυτούς τους χριστιανούς μάρτυρες και θα πρέπει να μην διαμαρτυρηθούμε. Όχι, σε καμία περίπτωση. Όσοι μαρτυρούν στην ε, Μέση Ανατολή και στην Αφρική ε, είναι περιπτώσεις που εντείνονται με την ανόητη πολιτική των ΗΠΑ και τις ε, παρεμβάσεις τους. Μιλώ για την παρέμβαση στο Ιράκ, στη Λιβύη, για την παρέμβαση στην Συρία, όπου λόγω αυτών των σχετικών παρεμβάσεων αυτή τη στιγμή θα ανατώνονται και σφάζονται οι χριστιανοί. Έχουμε το δικό μας μερίδιο ευθύνη πέραν α, της χαρακτηριστικής μας τοποθέτησης ως ευρωπαϊκής πολιτικής. Ε, ευχαριστούμε για 1,5 λεπτό ο κύριος Ντανζό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η επίθεση στο Κάρισα αυτά τα αποτρόπια εγκλήματα μας υπενθυμίζουν ότι η Ανατολική Αφρική όχι μόνο είναι περιοχή όπου υπάρχουν Ισλαμικές τρομοκρατικές επιθέσεις αλλά είναι και σημαντική αιστεία αποσταθεροποίησης Μέσω του Αλσαμπάμπ και της δράσης αυτών των τρομοκρατών στις διπλανές χώρες γίνονται παρόμοια, παρόμοιες επιθέσεις ε, με αυτά που κάνει το al η al στο Ισλαμικό Μαγκρέπ ή στη Μέση Ανατολή με το Ισλαμικό κράτος ή τον Μπόκο Χαράμ στην Κεντρική Αφρική. Το Al-Shabaab έχει χτυπήσει και άλλες χώρες, η τον μποκο χαραμ στην κεντρικη αφρικη το al εχει χτυπησει και αλλες χωρες η ουγγαντα για παράδειγμα και η Κένια φυσικά. Έχει υποστεί πριν από τον Καρύς άλλες επιθέσεις και στο Τζιμπουτί επίσης υπήρξαν ε, τρομοκρατικές απόπειρες. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε τι διαστάσει έχει αυτή η τρομοκρατική επιλή. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επανατονίσει τη στήριξή τη, που είναι σημαντική. Παρά όλα όσα υπονοούν ορισμένοι συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντική η στήριξη που δίνουμε στι αφρικανικέ δυνάμει στην περιοχή, στι χώρε ε, μεμονωμένα που αντιτίθεται στην τρομοκρατία. Δεν υπάρχει κανένα διαχωρισμό των θυμάτων τη τρομοκρατία. 150 φοιτητέ που δολοφονήθηκαν στην Κάρσα θυμίζουν του 150 που δολοφονήθηκαν στο Πεσάουα, στο Πακιστάν, το Δεκέμβριο του 2014. Δεν κάνουμε διακρίσει, αλλά πρέπει να σημειώσουμε παρόλα αυτά ότι οι τρομοκρατικέ ομάδες, οι Ισλαμικές, κυρίως ε, επιτίθενται στις ε, χριστιανικές μειονότητες παντού στον κόσμο. Και γι' αυτό η απάντησή μας πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις συμφωνίες με τις τρίτες χώρες που καταπολεμούν την τρομοκρατία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται πλήρως αυτές η, να συμπεριλαμβάνεται αυτή η διάσταση και να υπάρχει ένα είδος σύνδεσης της βοήθειας που δίνουμε στις χώρες αυτές με την καταπολέμηση της ε, Ισλαμιστικής τρομοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής ένα λεπτό, η Άννα Γκόμες. Η σφαγή στο Πανεπιστήμιο της Γκαρίσα δεν αξίζει απλώς την ε, έντονη αλληλεγγύη που θα πρέπει να εκφραστεί για τα θύματα αυτά και τον λαό της Κένιας. Η τρομοκρατία της Αλσαμπάμπ στην περιοχή παραμένει ατιμόρυτη και η κλιμάκωση των, εχθροπραξιών ε, απλώνεται και σε άλλε χώρε του κέρατο τη Αφρική. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τι κυβερνήσει τη Κένια και των γειτονικών χωρών να αναλάβουν τι ευθύνε του για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία και των ριζοσπαστικών ομάδων. Αγώνε όπου οι αναπτυξιακέ πολιτικέ έχουν ωφελήσει του λαού του και για τι οποίε θα πρέπει να δούμε ανταλλάγματα. Ε, στο Πανεπιστήμιο τη Γκαρίσα είχαμε ένα περιστατικό που δείχνει αλλαγή στάση και για την Κένια και για την περιοχή αυτή συνολικά. Η διεθνή κοινότητα λοιπόν θα πρέπει και αυτή να μεταβάλει τη στάση τη. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την παιδεία είναι θεμελιώδη δικαίωμα οποιασδήποτε κοινωνία θέλει να ονομάζεται δημοκρατική. Η Κένια και η Αφρικανική Ένωση θα πρέπει να δουν τι πραγματικέ ε, αιτίε του προβλήματο τη ριζοσπαστικοποίηση που ε, δίνουν τα επιχειρήματά του στου τρομοκράτε τη ομάδας Al-Shabaab που οδήγησαν στην θανάτωση 147 φοιτητών και άλλων ε, στην όλη περιοχή. Αν έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας. Ε, θα πρέπει να δώσουμε τέλος λοιπόν σε αυτήν την θεώρηση της τρομοκρατίας. Και πάλι να το πω σε αυτή τη συζήτηση για τελευταία φορά. Εάν έχετε ένα λεπτό για την ομάδα σας, δεν σας βοηθά να μιλάτε σαν πολυβόλο, διότι απλώς δεν μεταφράζεστε σωστά. Οπότε παρακαλώ προσπαθείτε να παραμένετε σε βασικά μηνύματα όταν έχετε λίγο χρόνο. Ή φροντίστε οι ομαδα σας να πάρουν περισσότερο χρόνο. Πάει ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη μια λοιπόν απέσια και απεχθή τρομοκρατική επίθεση αυτό το μήνα. Μια επίθεση εναντίον των νέων, εναντίον των φοιτητών, εναντίον των επαγγελματιών του μέλλοντος, των γονέων του μέλλοντος. Είναι ένας από τους στόχους λοιπόν των ομάδων τρομοκρατών να χρησιμοποιήσουν το πρόσχημα της ε, θρησκείας για να προκαλέσουν αναταράξεις. Και όποιος δεν ακολουθεί τα ίδια θρησκευτικά πιστεύω με αυτούς είναι άπιστος. Είναι άπιστος και πρέπει να καταστραφεί. Είδατε τι έγινε με τους Πακιστανούς οι οποίοι σχεδίαζαν μια επίθεση κατά του Βατικανού. Είδαμε τους δουλέμπορους που πέταξαν τους χριστιανούς στη θάλασσα πρόσφατα. Πρέπει λοιπόν τη μάχη κατά της τρομοκρατίας να την εντείνουμε, να είμαστε σε πιο στενή επαφή με τις αφρικανικές χώρες, την Αφρικανική Ένωση και να στηρίξουμε τις προσπάθειες που κάνουν στις χώρες αυτές για ειρήνευση. Θα είσαστε μοντέλο έτσι όπως μιλάτε για τους συναδέλφους σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, κύριος Ράνστορφ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Τσιγκίς Αϊτμάτοφ που ήταν συγγραφέα από το Κυργιστάν και μουσουλμάνος έγραψε ένα διήγημα. Ε, ε, Βασιζόμενο στην ιδέα πως το Ισλάμ δεν γνωρίζει τι σημαίνει άτομο. Και αυτό οδηγεί σε μια σύγκρουση μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών. Η Σαμπατίνα Τζέιμς είναι μια κυρία η οποία δεν δέχτηκε να παντρευτεί με προξενιό. Έγινε χριστιανή και την αντιμετώπισαν με εχθρότητα οι μουσουλμάνοι ομογενείς της. Και αυτό που, για το οποίο κατηγορεί την Ευρώπη είναι ότι είμαστε ανεκτικοί με τη μυσαλλοδοξία. Ναι, δεν μπορούμε εμείς να είμαστε ανεκτικοί με κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να ανεχόμαστε. Θα πρέπει να στηρίξουμε τους χριστιανούς και να τους προστατεύσουμε όπου στον κόσμο και να βρίσκονται. Ευχαριστώ Ιγνάτσιο Κορά, επίσης ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι, νομίζω όταν μιλάμε για 150 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους, είναι πολύ θλιβερό να βλέπουμε να μεταλλεύεται κανεί ε, την οποιαδήποτε ιδεολογία μπορεί να σχετίζεται με αυτό το θέμα. Είναι θλιβερό γιατί χρησιμοποιούμε τον όρο χριστιανή στο ψήφισμα, αλλά το θέμα είναι να αποδεχόμαστε δεν να αποδεχόμαστε ή όχι ότι ε, είναι χριστιανοί οι άνθρωποι αυτοί. Τα παιδιά αυτά ήταν χριστιανοί, είναι μειονότητα, εντάξει. Αλλά εάν ε, σταθούμε σε αυτό, είναι σαν να ε, επαναλαμβάνουμε το μήνυμα μίσου που είχε αποσταλεί εναντίον του στη χώρα του, στην Κένια. Και αυτό δεν είναι θετικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ενωμένη στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε μορφή τρομοκρατική επίθεση, είτε κατά τη χριστιανική μειονότητα, είτε οποιαδήποτε άλλη. Πολύ αποφασιστικά, χωρί να χρονοτριβεί. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το μήνυμα να βγει από αυτήν την ε, σύνοδο. Θα πρέπει να είμαστε πιο ενωμένοι στην αντιμετώπιση τέτοιου είδου φαινομένων. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ και εγώ. Α, έχει στηθεί μια μπλε ε, κάρτα. Ε, τη δέχεστε, η Τερέσα Χιμένα. Ναι, ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Κοράου. Ιγνάσιο, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αναφέρθηκε σε αυτά που είπες. Σε αυτά που είπα εγώ, ότι η αναφορά σε χριστιανούς δεν είναι ιδεολογικός πόλεμος. Αυτό που είπα εγώ είναι ότι στο ψήφισμα που θα υποβάλουμε, ο τίτλος του ψηφίσματος, εκτός από την γένεια, είναι η διώξεις των χριστιανών. Εάν δεν αναφέρετε στο ψήφισμά σας παρά μόνο δύο φορές τους χριστιανούς, κάτι δεν, δεν πάει καλά. Αν κάνουμε ένα ψήφισμα για τις διώξεις στους ε, ε, Ρωμά, για παράδειγμα, και στο εσωτερικό του ψηφίσματος δεν αναφέρουμε τους Ρωμά, άρα κάτι κάνουμε λάθος. Αυτό είναι το μόνο που θέλω να τονίσω. Πρόεδρος. Η διαδικασία της μπλε κάρτας είναι για να κάνετε ερωτήσεις στους ομιλητές όχι για να ε, διορθώσετε θέματα με τα οποία διαφωνείτε στην ομιλία τους. Δεν ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε σε κάποια ερώτηση. Εντάξει, συμφωνώ με τη συνάδελφο Χιμένεθ. Α, είναι σωστό και δίκαιο να καταδικάσουμε μια επίθεση κατά της χριστιανικής μειονότητας. Όντως, υπερασπιζόμαστε τα θεμέλια της Ευρώπης, την ε, ιστορία της, την χριστιανική της καταγωγή. Αυτό που έλεγα απλώς είναι ότι στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των διαφορών ομάδων δεν θα πρέπει να στεκόμαστε στα λόγια, στους όρους, διότι το μήνυμα που προκύπτει είναι αναρνητικό για κάτι που είναι τόσο σημαντικό και ένα ε, πρόβλημα που έχει πάρει διεθνείς διαστάσεις. Δεν αφορά μόνο το Shabaab, αλλά το Ισλαμικό κράτος, το Ίζης, το Μπόκο, το Χαράμ. Εδώ μιλάμε Μιλάμε λοιπόν για ένα σωρό μειονότητε που απειλούνται. Αυτό ήταν το νόημα τη παρέμβασή μου. Τώρα ο λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το τραγικό και κατακριτέο περιστατικό της ε, δολοφονίας των 147 φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Γκαρίσα της Κένια έφερε στην επιφάνεια μια πραγματικότητα στην οποία δυστυχώς δεν είχαμε δώσει μέχρι τώρα τη δέουσα σημασία πρόκειται για τις δολοφονίες των χριστιανών παγκοσμίω από εξτρεμιστικές ισλαμιστικές οργανώσεις. Ε, σε έκθεση της ε, οργανώσεως open doors αναφέρεται ότι από τα 50 κράτη που διώκουν σήμερα τους χριστιανούς τα 40 είναι μουσουλμανικά. Δηλαδή το 80% των χριστιανών διώκεται από μουσουλμάνους κάθε πολιτικής τοποθετήσεως. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο και δεν πρέπει να μα προκαλεί έκπληξη το γεγονό ότι οι χριστιανοί στοχοποιούνται από ακραίου Ισλαμιστέ, τρομοκράτε δυστυχώ αυτή την κατάσταση την έχει υποθάλψει και την συντηρεί η αδιαφορία των χωρών τη ίσο και κυρίω τη ευρωπαϊκή ενώσεω. πιο πολύ ενδιαφερόμαστε για την παραβίαση των δικαιωμάτων των τρομοκρατών και όχι για την προστασία τη ζωή των θυμάτων του. ουδή πέραν του θεού έχει το δικαίωμα να αποφασίσει πότε θα πεθάνουμε πού θα πεθάνουμε και πόσα θα ζήσουμε. γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αντιδράσουμε να οργανωθούμε και να Αντιμετωπίσουμε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. διαφορετικά θα θρηνήσουμε θύματα. η υπομονή και η ανοχή μας έχουν όρια τα οποία πλέον έχουν εξαντληθεί. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, για άλλη μια φορά εδώ ε, κλαίμε για νεκρούς αλλά και θρυνούμε αλλά δεν έχουμε το θάρρος να πούμε ότι έχασαν τη ζωή τους γιατί εμείς δεν έχουμε το θάρρος ή είμαστε δειλοί ή μας φοβίζει κάτι που εξαπλώνεται σε όλη μας την Ήπειρο, η χριστιανοφοβία δηλαδή. Εδώ λέμε πράγματα που δεν ε, κολλάνε πουθενά. Θα πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει κάποια ευθύνη. Λέμε ότι εμείς προσπιζόμαστε τα δικαιώματα. Μα πώς προσπιζόμαστε τα δικά μας θεμελιώδη δικαιώματα. Η ανεξιθρησκεία είναι το πλέον ε, ιερό από τα δικαιώματα. Είναι αυτό από το οποίο εκπορεύονται όλα τα υπόλοιπα. Ε, δεν μπορούμε μπορούμε να ξεχνάμε ότι η ανεξαρτησία και το επίπεδο ελευθερία είναι αλληλένδετα. Ε, έχουμε τον Πάπα, ο οποίο λέει ότι η αδικία πρέπει να καταδικάζεται και να ε, εξαλείφεται. Πώ τον χειροκροτούμε. Ε, πραγματικά είμαι τελείω ε, ευνηδιασμένη όταν μιλάμε για την Κένια και λέμε ότι οι χριστιανοί είναι μειονότητα. Μα ε, οι χριστιανοί στην Κένια είναι το 83% του πληθυσμού. Οπότε οι χριστιανοί είναι μάρτυρε ε, όταν είναι μειονότητα αλλά και όταν είναι πλειοψηφία. Ε, τον περασμένο αιώνα είχαμε τον αιώνα ε, των χριστιανών μαρτύρων περισσότερο και από ό,τι στι διώξει τη αρχαία Ρώμη. Ε, Στου διωγμού. Εδώ λοιπόν έχουμε τραυματικά γεγονότα, άνθρωποι που καίγονται, τους καίνε στην πυρά ε, και άλλα. Ε, πρέπει να έχουμε την τόλμη να πούμε είμαι χριστιανός πλέον. Ευχαριστώ πολύ. Δέχεστε μια μπλε κάρτα παρακαλώ από τον κύριο Κοράου. Ωραία. Παρακαλώ. Ο κύριος Κοράου. Ευχαριστώ Ήθελε να σε ρωτήσω τη συνάδελφο Γκαρντίνη. Στην Κένια θανατώθηκαν μη μουσουλμάνοι. Δεν ήταν η επίθεση ιδιαίτερως κατά των χριστιανών. Σας το ζητώ αυτό λοιπόν και σας παρακαλώ, εάν εμείς ως κοινοβούλιο τοποθετηθούμε για να μιλήσουμε για πλειοψηφία χριστιανών ή μειοψηφία χριστιανών, ε, παρα, παραποιούμε τα γεγονότα. Βεβαίω, να καταδικάσουμε οποιαδήποτε επίθεση λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων. Γκαρντίνη, συμφωνώ απολύτω. Γι' αυτό για το βραβείο Ζαχάροφ είχα προτείνει τον Πατριάρχη του Ιράκ. Διότι πρόκειται για μια προσωπικότητα που υπερασπίζεται όλε τι χριστιανικέ μειονότητε που ζουν στο Ιράκ. Όταν όμω μιλάμε για μια σφαγή τέτοιων διαστάσεων, όταν τα πρόσωπα επιλέγονται βάσει των θρησκευτικών του πεπιθήσεων και θανατώνονται διότι δεν ε, σέβονται το Κοράνι ή γιατί έχουν ένα σταυρό πάνω του, μιλάμε για μάρτυρε χριστιανού και είναι πάρα πολλοί και είναι πολυαριθμότατοι λοιπόν οι χριστιανοί που έχουν μαρτυρήσει δεν πρέπει να έχουμε τη δηλία να ε, αναγνωρίζουμε την πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Επόμενη μιλήτρια για ένα λεπτό η Νίνα Γκύρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στοχεύοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την εκπαίδευση όπω τόσο πρόσφατα στο Γκαρίσα στην Κένια, επιτιθέμενη κατά τη UNICEF, το προσωπικό όπω την προηγούμενη εβδομάδα στη Σομαλία, η Al Shabaab βάζει βόμβα κάτω από το μέλλον τη Αφρικανική Υπήρου. Σίγουρα δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Είναι απόλυτα απαράδεκτο και τα συλληπιτήριά μου στι οικογένειε ε, των θυμάτων και που το μέλος των οικογενειών τους ε, καταστράφηκε και οι επιπτώσεις τη δράση αυτών των οργανώσεων στι διάφορες χώρες και το παγκόσμιο ανεπτυγμένο σύστημα χρηματοδότησή τη σε συνδυασμό με άλλες τρομοκρατικές οργανώσει, σημαίνουν ότι χρειάζεται ευφυή, αποτελεσματική και συνολική αντίδραση. Και γι' αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε και να συντονίσουμε τη δράση μας με την ε, κυβέρνηση τη Κένια, που ναι μεν καθυστέρησε να αντιδράσει και καθυστέρησε με τρόπο πολύ περιορισμένο. Οποιαδήποτε στρατηγική και αν υιοθετήσουμε θα πρέπει να λύσει και όχι να συμβάλλει στις διαιρέσει που προσπαθεί να υποθάλψει αυτή η οργάνωση. Και πιστεύω ότι οποτεδήποτε μία εθνότητα, μία ομάδα του πληθυσμού διώκεται, όλη η κοινωνία πλήγεται και να έχουμε υπόψη μας ότι οι δραστηριότητες αυτές στην Κένια έχουν περιθεροποιήσει και ε, στιγματίσει και μουσουλμανικές ε, μειονότητες. Άρα χρειαζόμαστε μια στρατηγική μαζί με την κυβέρνηση που να σημαίνει ασφάλεια για όλους ανεξάρτητα από τη θρησκεία ή την ομάδα στην οποία ανήκουν. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής ε, για ένα λεπτό, Φραντς Ομπεμάερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. 147 φοιτητέ δολοφονήθηκαν από αυτήν την Ισλαμιστική οργάνωση. Σύμφωνα με τις ε, δικές της, ε, με τα δικά της, ε, με τις δικές της δηλώσεις ήθελαν να δολοφονήσουν χριστιανούς και αν δεν το εμποδίσουμε αυτό δεν, δεν κάνουμε το καθήκον μας. Πρέπει να υποστηρίξουμε την Αφρικανική Ένωση για να αντιμετωπιστεί η Al Shabaab και στη χώρα προέλευσης, στην Σομαλία. Χρειάζεται αποφασιστική δράση. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, αλλά θα έπρεπε να έχουμε το θάρρος να βάλουμε το σημείο αυτό και στον τίτλο του κειμένου, ότι είναι Ισλαμιστική βία. Πρέπει να αναφέρουμε λοιπόν ότι οι χριστιανοί διώκονται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο διωγμός των χριστιανών δεν προέρχεται από ναζί, από κομμουνιστές, από βουδιστές, αλλά από το επιθετικό ακραίο Ισλάμ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ομπερμάιο. Για 1,5 λεπτό ο συνάδελφος Ντάβος Στήρ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας ε, τα συλληπιτήριά μου ε, στις οικογένειες των θυμάτων στην Κένια. Αν βασιστούμε στους αυτόπτες μάρτυρες, ε, στοχοποιήθηκαν οι φοιτητέ που ήταν χριστιανοί. Αυτό δεν αποτελεί όμως ε, δυστυχώς εξαίρεση. Το 70% των χριστιανών του Ιράκ χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι χριστιανοί στη Συρία έχουν μειωθεί αριθμητικά εξίσου Οι χριστιανοί λοιπόν είναι η ομάδα που διώκεται πιο πολύ λόγω χριστιανικών πεπιθήσεων. Κάποιοι δεν το δέχονται. Είναι όμως ε, εκπληκτικό μη μυσαλλοδοξία αντιμετωπίζουμε από πάρα πολλούς ευρωβουλευτές όταν συζητάμε το θέμα αυτό. Προφανώς μπορούμε να μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα, αλλά δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε για διωγμό χριστιανών. Και δεν μιλάμε μόνο για διωγμό. Φαίνεται πως δεν μας επιτρέπεται να αναφερόμαστε καν στη θρησκεία, παρόλο που αποτελεί κομμάτι της, της ζωής μας και δεν αποτελεί μόνο κομμάτι της ε, ιδιωτικής μας ζωής, αλλά έχει και μια κοινωνική διάσταση, μια τέτοια προσέγγιση τόσο φανατική, όντως προκαλεί ε, ακραίες αντιδράσεις, που τελικά ίσως οδηγήσουν στο τέλος της Ευρώπης με τη μορφή που τη γνωρίζουμε. Για το λόγο αυτό χρειάζεται διάλογος. Και πρέπει να σας πω ότι αντιμετωπίσαμε και μια προσπάθεια να μην εγκριθεί το ψήφισμα για το σχετικό θέμα δεν θα παραιτηθούμε. Θα συνεχίσουμε να υψώνουμε τη φωνή κατά ε, των φανατισμών και των διωγμών των χριστιανών. Καλησπέρα σας συνάδελφοι, ευχαριστώ. Η ε, κυρία Μίζη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Παρά το γεγονός ότι η ανεξιθρησκεία είναι ένα θεμελιώδες ε, δικαίωμα, Φαίνεται ότι είναι μια αρχή η οποία δεν διασφαλίζεται παντού. Η Κένια είναι μια χώρα με πολιτιστικέ και θρησκευτικέ ε, και κοινωνικέ διαφορέ. Δυστυχώ όμω υπάρχει και φοβερή ανισότητα και υπάρχει και ριζοσπαστικοποίηση στι θρησκευτικέ πεπιθήσει. Φαίνεται εδώ να καταπιέζονται τα δικαιώματα των ε, πολιτών τη Κένια, οι οποίοι θέλουν να ζήσουν ειρηνικά και ελεύθερα. Εδώ ε, φαίνεται να μην προστατεύεται το θεμελιώδε δικαίωμα τη ελευθερία. Πρέπει να βρούμε καλύτερε λύσει για την καταπολέμηση κάθε μορφή τρομοκρατία και να προστατεύουμε την, ε, ε, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τέτοιου επιθέσει. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι προστατεύουμε τους φοιτητέ και τους ενθαρρύνουμε να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Πρέπει να ε, βεβαιωθούμε ότι ο κάθε λαός έχει δικαίωμα στην ε, παιδεία και στην ανεξιθρησκεία. Η Αφρικανική Ένωση μαζί με τη Διεθνή Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσουν τις διαρκείς και συγκεκριμένες λύσεις που χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν αυτές τις τρομοκρατικές ομάδες και να βρουν και διαρκείς λύσεις για την ειρήνευση και την σταθερότητα στην περιοχή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κυρία Μίτζη ε, που σεβαστήκατε το χρόνο Δέχεστε γαλάζια κάρτα από τον κύριο Νέκοφ. Κυρία Μίτζη. Κύριε Σενέκοφ. 30 δευτερόλεπτα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Στο κέρας της Αφρικής έχουμε μια περιοχή η οποία γίνεται όλο και πιο ακραία. Δεν υπάρχει σταθερότητα και από εκεί προέρχονται κύματα μεταναστών. Τι πιστεύετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένα μέτρα? στη μάχη κατά του προβλήματος αυτού. Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε μια στρατηγική η οποία να μας ικανοποιεί όλους και το κάνουμε χρόνια τώρα. Πρέπει να σας πω πως ε, στο κέρας Αφρικής ε, έχουμε πολλές εθνότητες, πολλούς πολιτισμούς και μερικά από τα προβλήματα είναι οικονομικής φύσης. Υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα τρομοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να τους θεωρεί όλους ίδιους και δεν μπορεί να προσφέρει σε όλους παρόμοιες λύσεις. Είναι διαφορετικά τα προβλήματα. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει πως οι λύσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν σε κάθε μεμονωμένη χώρα. Κυρία Αλιωμαρή, για ένα λεπτό. Ενάμιση λεπτό. Ο λόγος είναι σε εσά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν το κατάλαβα. Νομίζω είναι απαραίτητο, όπως είπαμε σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δεν μπορούμε να λέμε συγχρόνως, και αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα, πως η Ευρώπη βασίζεται σε χριστιανικά θεμέλια και από την άλλη να μην δείχνουμε ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Πρόκειται για ένα πραγματικό γεωστρατηγικό πρόβλημα. Σήμερα υπάρχει βούληση από κάποιες ομάδες να δημιουργήσουν μία κάποια ομαδοποίηση θρησκευτική σε κάποια κράτη και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Από τη στιγμή που θα έχουμε μόνο θρησκευτικά κράτη θα αντιμετωπίζουμε προβλήματα και εντάσεις μεταξύ αυτών και των όμορων κρατών. Και έτσι θα γενικευθεί ο πόλεμος και τα όσα παίζονται. Είναι θέμα γεωστρατηγικής λοιπόν. Έχουμε πρόβλημα και φιλοσοφικής φύσης και παράλληλα έχουμε και πρόβλημα πολιτικό-ανθρωπιστικό. Η Ευρώπη λοιπόν που θέλει να θεωρείται ε, η υποστηρή που στηρίζει την αδελφότητα μεταξύ των λαών και την ανεκτικότητα να ε, επιβάλλει την αναγνώριση των δικαιωμάτων όλων. Γιατί για τους χριστιανούς της Κένια έχουμε ευθύνη και γενικότερα θα πρέπει να σταθούμε υπεύθυνοι για όλους τους χριστιανούς που είναι μειονότητες που διώκονται να τους στηρίξουμε, να τους στηρίξουμε όχι μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις. Το να είναι κανείς ε, βουλευτής δεν είναι μόνο, να, δεν είναι ε, μόνο ωραίοι λόγοι, αλλά είναι και πράξεις. Λοιπόν, ο κύριος Νεγκρέσκου σας ε, σηκώνει γαλάζια κάρτα, θα διδεχτείτε. Σας άκουσα με πολύ προσοχή, ήσασταν υπουργό στη Γαλλία και σας ρωτώ το εξής δηλαδή, δράση θα θέλατε να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση γιατί μιλήσατε για ε, μόνο θρησκευτικά κράτη Ακριβώ ε, λοιπόν, προτείνεται για αυτό στρατιωτική δράση, ανθρωπιστική δράση. Πώ μπορούμε να αποφύγουμε πω τέτοιου είδου γεγονότα θα επαναληφθούν στι χώρε αυτέ. Νομίζω πω έχουμε δύο-τρία είδη δράση που θα μπορούσαμε να αναλάβουμε. Πρώτα απ' όλα σε επίπεδο διακυβερνητικό. Προφανώ δεν μπορούμε εμεί να υποκαταστήσουμε τι κυβερνήσει αυτών των χωρών. Αντίθετα όμως υπάρχει υποχρέωση διαλόγου, συζήτησης, στεναρής συζήτησης, για να τους δείξουμε πως δεν είναι προ συμφέρον τους ένα τέτοιο είδου σύστημα μια θρησκεία να εγκαθιδρυθεί στη χώρα του. Επίση, έχουμε την υποχρέωση και το καθήκον τη πεποίθηση, τη πειθού, με συγχωρείτε, αλλά και τη εκπαίδευση να του δείξουμε τι σημαίνει ανοχή και ανεκτικότητα. Ευχαριστώ για ένα λεπτό, κύριο Σπαρνιό, ε, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, ο τρόμος είναι αυτό που ζήσαμε στις αρχές Απριλίου με την ε, δολοφονία 147 φοιτητών από την ομάδα ε, Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί οι διοικητικές αρχές της Κένιας παρέμεναν αδρανείς ενώ ο τύπος ήταν ήδη παρόν. Γιατί πέρασαν τόσες ώρες μέχρι ο στρατός της Κένιας να παρέμβει. Πρόκειται για ένα ερώτημα ε, πολύ χειροπιαστό και πραγματικά νομίζω ότι πρωτεύει να θέσουμε τα σωστά ερωτήματα ω ε, ευρωβουλευτέ. Μα έχει απασχολήσει ήδη η ασφάλεια στην ε, περιοχή αυτή. Ήδη υπό την ηγεσία του κυρίου Πέτρη είχαμε επισκεφτεί την Κένια για, στα πλαίσια τη κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα και τη Σομαλία. Κύριε Επίτροπε, δεν πιστεύετε ότι χρειάζεται μια στρατηγική για την περιοχή αυτή, για το κέρα τη Αφρική. Δεν πρέπει να δούμε την εντολή τη επιχείρηση επιχειρήσεις ε, ITM στην Σομαλία για να καταπολεμήσει γενικότερα τι δημοκρατικέ ομάδες της περιοχή Πρόεδρος, ευχαριστούμε ο κύριο Κέλλερ για ένα λεπτό. Στην Κερίσα σχεδόν 150 αθώοι νέοι δολοφονήθηκαν. Οι περισσότεροι ήταν χριστιανοί. Τους ξεχώρισαν από τους άλλους και τους δολοφόνησαν. Η καταγγελία και οι εκφράσεις αλληλεγγύης είναι αναγκαίες αλλά όχι επαρκείς. Στην Καρίσα υπήρχαν δεκαπλάσια αθώα θύματα από αυτούς που δολοφονήθηκαν στο Σαγλί Εμπτό και την άλλη επίθεση στο Παρίσι. Δεν είναι θέμα αριθμών, είναι θέμα αντίδραση με την ίδια αποφασιστικότητα. Πρέπει λοιπόν όλοι σήμερα να δηλώσουμε, όπως είπε η συνάδελφος Γκαρντίνη, και εγώ είμαι χριστιανός για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διώξη των χριστιανών, για τη μετώπιση δηλαδή της ε, διώξη των χριστιανών, πρέπει να είναι στοιχείο τη στρατηγική μας για τις σχέσεις μας με τρίτες χώρες και για τις άλλες θρησκείε. Πρέπει να καλέσουμε τους ε, μουσουλμάνους ηγέτες να να ακολουθήσουμε το αποτέλεσμα, να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του βασιά της Ιορδανίας που είπε ότι όλες οι επιθέσεις είναι επιθέσεις κατά της ε, μουσουμανικής θρησκείας. Η κυρία Τζούφρεντα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η σφαγή των χριστιανών φοιτητών στην Κένια προκαλεί την καταδίκη και την, τον αποτροπιασμό και πάλι για λόγους ε, πολιτιστικούς ε, για, κατά τις γνώσεις έντρασαν τρομοκρατικές ομάδες. Η οργή, η δολοφονική οργή του εξτρεμισμού των ε, Ισλαμιστών οδηγεί και σε ένα άλλο παράδεκτο φαινόμενο. Εδώ χτυπήθηκε ένα πανεπιστήμιο, το ίδιο το σύμβολο της ειρηνικής συμβίωσης και της αμοιβαίας συνεννόησης. Εδώ ε, φαίνεται να θέλουν να διαγράψουν το μέλλον, να υποδουλώσουν τους νέους που να είναι υποχείρια του τρόμου και της έλλειψης γνώσης και της ε, έλλειψης φαντασίας. Οι τρομοκράτες έχουν τον εξή λόγο. Οι νέοι σπουδάζοντα ε, μπορούν να χειραφετηθούν, μπορούν να οικοδομήσουν ένα μέλλον ελευθερίας, μπορούν να συλλογιστούν και να σκεφτούν μια νέα τάξη πραγμάτων. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη αυτή την ελπίδα κυρίως να τους εξασφαλίσει, να στηρίξει, να στηρίξει τους φοιτητές για να μην ξαναγίνουν ποτέ θύματα της βίας. Ευχαριστώ κύριο Τόκιος. Ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το ψήφισμά μας σήμερα καταδικάζει, όλοι μας καταδικάζουμε από κοινού τις ε, διώξεις και τις επιθέσεις κατά των χριστιανών παντού στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένες στις κτηνόδους δολοφονίες των φοιτητών στην Κένια. Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να είμαστε ενωμένοι έναντι όλων των παραβιάσεων τη της ε, θρησκευτική συνείδηση και άλλων πεπιθήσεων γιατί είναι θεμελιώδη δικαίωμα. Οι χριστιανικές ρίζες της Ευρώπης απαιτούν να είμαι θα υπεύθυνοι για τους χριστιανούς παντού στον κόσμο. Οι χριστιανοί είναι η πιο διοκόμενη θρησκευτική ομάδα στον κόσμο. Η Αλσοβά που δημόσια δηλώνει ότι κάνει πόλεμο κατά των χριστιανών με βάση τη σημερινή μας απόφαση ας ε, αποφασίσουμε ότι η διώξη κατά των χριστιανών είναι προτεραιότητα για την Ένωση για όλους μας και για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και για την Ένωση και για τα κράτη-μέλη. προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ζωής είναι καθήκον μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάιντιν Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αυτά τα φρικτά γεγονότα στην Καρίσα δεν είναι μεμονωμένα. Είναι κάτι που συμβαίνει σχετικά τακτικά. Υπάρχει κάποιο πρότυπο. Το Ισλάμ, ορισμένοι μουσουλμάνοι επιτίθενται κατά των χριστιανών, άλλων ε, μειονοτήτων και κατά των γυναικών. Όπως και τον Μπόκο Χαράμ, όπως και τον Ντάες. Όλοι αυτοί επιτίθενται κατά των ίδιων ομάδων. Γίνονται καταστροφές, καταστροφές αυτών που θεωρούμε ιερά και κατόπιν ε, δημιουργείται ένα τρομοκρατικό καθεστώς. Χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση γιατί πίστευα ότι πολύ σύντομα θα εξαφανίζονταν ε, τα νέα αυτά από τον κόσμο γιατί υπάρχει κάποιο είδους ιεράρχηση αυτών των ε, γεγονότων, αυτών των θηριωδιών αλλά οι ανθρώπινες ζωές είναι πάντα ανθρώπινες ζωές για οποιοδήποτε λόγο και αν συμβαίνουν και πρέπει να τις καταδικάζουμε. Τις ε, ε εναντίον τους. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό κύριο Σαντάκτουσον. Ευχαριστώ πολύ. Ένα από τα θύματα που επιβίωσε της επίθεσης ε, στην Καρίσα μας είπε τα εξής. Οι φοιτητές, οι χριστιανοί χωρίστηκαν από τους ε, μουσουλμάνους και όσοι ήταν χριστιανοί δολοφονήθηκαν αμέσως. 147 αθώες ζωές χάθηκαν. Αρκετοί αποκεφαλίστηκαν και την ώρα που τους αποκεφάλιζαν οι δράστες εκφωνούσαν το Κοράνι. Τέτοιες επιθέσεις κατά χριστιανών έχουμε πάρα πολύ στον κόσμο. 300 εκατομμύρια χριστιανοί κινδυνεύουν και εκατοντάδες χιλιάδες κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους επειδή πιστεύουν στον χριστιανισμό. Έχουν χαθεί οι χριστιανικοί πληθυσμοί στις μουσουλμανικές χώρες γιατί οι Ισλαμικές δυνάμεις προχωρούν. Έχουμε καθήκον να δράσουμε. Αντιμετωπίζοντας τέτοια φαινόμενα θα πρέπει ε, στο βορρά της ε, χώρας αυτής να δημιουργήσουμε ε, μια ζώνη ειρήνης για να μην διώκονται οι χριστιανοί. Επόμενος ο μιλητής είναι ο κύριος Χέτινα που είναι και τελευταίος μας ο μιλητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ κυρία Πρόεδρε να μιλήσω για το ολοκαύτωμα το οποίο αποτελεί ένα παράδειγμα συλλογικής ενοχής. Έχουμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε το 1915 την περίπτωση της Τουρκίας με τους Αρμενίους. Οι Τσετσένοι λένε πως το μόνο λάθος που έχουν κάνει είναι που γεννήθηκαν Τσετσένοι, γιατί 80.000 δολοφονήθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις. Οι Χούτου δολοφονούσαν Τούτσι στη Ρουάντα και η συλλογική ενοχή κρύβεται πίσω από τα γεγονότα στην Γκαρίσα η αντιχριστιανική, το αντιχριστιανικό μίσος, ε, τα γεγονότα στην Τσάρλι ε, Επτό, αυτές οι εχθρότητες, η χριστιανοφοβία, η ισλαμοφοβία είναι φαινόμενα τα οποία τρέφουν το ένα το άλλο. Και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει ειρήνη μεταξύ των θρησκειών, δεν θα βασιλεύσει η ειρήνη στον κόσμο. Περνάμε στη διαδικασία προσέλκυση τη προσοχή του προέλθου. Έξι θα πάρουν το λόγο και θα σεβαστούμε φυσικά την, το σχετισμό δυνάμεων. Ο κύριος, Πέτερ, ο κύριος Πρέτσεν, η κυρία Πρέτσεν. Ευχαριστώ. Οι μεγαλύτερε διώξει χριστιανών στον κόσμο συμβαίνουν στη Βόρεια Κορέα, τη Σομαλία, το Ιράκ, τη Συρία και το Αφγανιστάν. Οι χριστιανοί διώκονται, ε, ασκείται βία εναντίον του. Στην ε, Βόρεια Κορέα, την Σομαλία και το Ιρακό. όχι μόνο απαγορεύεται να ασκεί κοντά ακόμη και να σκέφτεσαι για τη θρησκεία είναι επικίνδυνο. Αν υπάρχει παραμικρή υποψία ότι είναι πιστή σε μια θρησκεία, ακόμη και αν δεν εκτελούν θρησκευτικά καθήκοντα, εκτελούνται. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τέτοιε παραβάσει των πέντε δικαιωμάτων. Πρέπει να πούμε την αλήθεια. Πρόκειται για γενοκτονία σε τέσσερι υπήρου. Οι δολοφονίε ε, των φοιτητών στην Κένια είναι συνέχεια αυτών που βλέπουμε στο Πακιστάν, την Ιγυρία. Εάν κάποιο δολοφονεί φοιτητέ επειδή είναι χριστιανοί, δολοφονεί το μέλλον μια θρησκεία. Την, η παλιότερη θρησκεία στον κόσμο, η οποία έχει επιβιώσει ε, εδώ και 2.000 χρόνια παρά τι διώξει, Πόσο καιρό θα αγνοούμε αυτή την κατάσταση και θα νύπτουμε τα σχήρα μα όπω ο πόντιο πιλάτο. Πιστεύω ότι πρέπει να πούμε ότι αρκεί. Ο κύριο Καπούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η θρησκεία σε πολλά μέρη του κόσμου κινδυνεύει. Διωγμή κατά των χριστιανών που πολλαπλασιάζονται, βία από ένοπλες ομάδες και παράνομους τρομοκράτες. Οι χριστιανοί είναι θύματα αιματηρών επιθέσεων από τη Μέση Ανατολή στην Ινδία, από την Αφρική στο Πακιστάν. Δεν αρκούν οι κλήσεις του Πάπα Φραγκίσκου προ την διεθνή κοινότητα. Παραμένουμε αδρανείς μπροστά στι σφαγέ αυτέ. Σήμερα σε σχέση με το παρελθόν βλέπουμε να υπάρχουν εντονότεροι, μεθοδικότεροι και ε, ιδεολογικοί διωγμοί. Οι χριστιανοί είναι στόχο διωγμών είτε από εξτρεμιστέ του Ισλάμ γιατί γίνονται αντιληπτοί ως κίνδυνος για το Ισλάμ είτε γιατί είναι εμπόδιο στι χώρε τη Μεσανατολή για να εξασκήσουν ε, τι πολιτικέ του οι Ισλάμιστέ που είναι ακραίοι. Η σφαγή στην Κένια... Ε, διαπράχθηκε από ε, μια ομάδα που ε, μπήκε σε ένα πανεπιστήμιο παραβιάζοντας τις πύλες ε, και οδήγησε το θάνατο 147 φοιτητών. Θα πρέπει να λάβουμε το μέρος διευθύνη μας και η Ευρώπη να καταστρώσει τη σωστή πολιτική. Ευχαριστώ, αλλά θα ήθελα να σας πω να μιλάτε πιο αργά, αλλά ε, Ο Κύριος Μαριάς, ένα λεπτό. συναλλαγές κατά των χριστιανών σε διάφορα μέρη του κόσμου δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. τελευταίο κρούσμα η αποτρόπαια σφαγή 147 χριστιανών φοιτητών στην πανεπιστημιούπολη της γκαρίσα στην κένια από την αλ σαμπάμπ που έχει τη βάση της στη σομαλία. οι τζιχαντιστές του ίσις της μπόκο χαράμ της αλ σαμπάμπ εντείνουν τις επιθέσεις τους κατά των χριστιανών στη συρία τη λιβύη την κένια την νιγηρία και σε άλλα μέρη του κόσμου βεβαίως οι τζιχαντιστές δρούν και κατά των μουσουλμάνων στις διάφορες αραβικές χώρες. οι τζιχαντιστές προσπαθούν να προκαλέσουν θρησκευτικούς πολέμους που όπως γνωρίζουμε ιστορικά ήταν ιδιαίτερα αιματηροί. όμως τα αίτια των συγκρούσεων στην κένια και στο κέρας της αφρικής δεν έχουν θρησκευτική βάση. οφείλονται στη φτώχεια την αρπαγή των γεών στην υπερεκμετάλλευση χριστιανών και μουσουλμάνων από τα διάφορα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα διερωτώ με άραγε αν η θεωρία της σύγκρουσης των πολιτισμών που αναπτύχθηκε πριν μερικές δεκαετίες ήταν μια πρόβλεψη ή μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάκοφσιτς, ένα λεπτό επίσης. η μια αυτοεκπληρουμενη προφητεια ευχαριστω ευχαριστω ο κυριος ενα λεπτο επισης Αλσαβάμπ είναι μόνο μία από τις τρομοκρατικές οργανώσεις που τρομοκρατούν τους λαούς μας, τους λαούς του κόσμου. Και όπως όλες οι τρομοκρατικές οργανώσεις, επιλέγει τα θύματά της και τους στόχους της πολύ προσεκτικά. Προσεκτικά λοιπόν έτσι επέλεξε και το, την Πανεπιστημίου της ε, Γκαρίσα για να δολοφονήσει νέους. Για να δολοφονήσει το μέλλον ε, μιας ολόκληρης χώρας μέσω αυτών των δολοφονιών για να μπορέσει να στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι η δύναμη της βίας ε, θα κυριαρχήσει. Αλλά εμείς ε, πρέπει να αντιταχθούμε. Να αντιταχθούμε στη θεωρία της σύγκρουσης των πολιτισμών, να αντιταχθούμε σε θρησκευτικούς πολέμους. Αυτό είναι το μήνυμά μας και είμαι βέβαιος στο Κοινοβούλιο θα στέλνει ένα τέτοιο μήνυμα. Ευχαριστώ κύριο Πόλτσακ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αναρωτιόμουν αν είχε έννοια να πάρω τον λόγο. Και παίρνοντας το λόγο, θα ήθελα να αναλογιστούμε όλοι τι λένε τα θύματα για αυτά που λέμε εμείς εδώ. Νομίζω ότι θεωρούν ότι είναι γελίες οι διακηρύξεις μας. Ο Πάπας και θρησκευτικοί ηγέτες του Ισλάμ καταδίκασαν αυτές τις πράξεις τονίζοντας ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτούς που ριζοσπαστικοποιούνται και τόνισαν ότι μαζί ως χριστιανοί και ως μουσουλμάνοι ηγέτες καταδικάζουν αυτές τις μεθόδους. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε μια κοινή δήλωση που να λέει ότι η θρησκευτική βία θα ριζοσπαστικοποιήσει ε, πολλές νέες γενιές. Ο κύριος Φουντσούλικα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ να μιλήσω την ε, να μιλήσω τελευταίως. Τα, η ζωή ε, ανθρώπων έχουν χαθεί λόγω της φτώχειας, της περιφερειοποίησης και αυτό μας οδηγεί σε δράματα όπως αυτό της Γκαρίσα φαίνεται την τελευταία δεκαετία. Τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον σχολών, πανεπιστημίων και ιδρυμάτων έχουν απολαπλασιαστεί μέσα στα πλαίσια της διεθνούς τρομοκρατίας. Αυτό δεν είναι απλώς σύμπτωση. Ε, οι τρομοκράτες μισούν την παιδεία και την μάθηση, διότι κάποιοι ε, πιθανώς αποκλείστηκαν από ε, αυτή την ε, Αυτή είναι ε, μια απόδειξη για το ότι μπορούμε να καταπολεμήσουμε τα αίτια της τρομοκρατίας, τι εξτρεματικές αυτές ομάδες που επιτίθενται σε νέου πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και ε, η πανάπτυξη, η έλλειψη δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, θεσμικά, οικονομικά και κοινωνικά, ε, διακριτικέ μεταχειρήσει ε, κατά των μειονοτήτων, ε, συστηματικέ παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι αυτά που οδηγούν τι ομάδε των εξτρεμιστών να ε, δρουν έτσι λόγω φτώχεια και τη γενικευμένου αισθήματο ανασφάλεια. Σα ευχαριστούμε. Δεν ήσασταν ακριβώ ο τελευταίο. Ο κύριος Κέμ. Πρόεδρε, Πρέπει να καταδικαστεί ο εξτρεμισμός οποιαδήποτε και ιδεολογία αν τον υποθάλπη είτε οποιοδήποτε πολιτικό πρόσχημα. Η ομαδα al Αλ-Σαμπάμπ, το Ισλαμικό κράτο, η Al-Qaeda είναι ομάδες που πρέπει να καταδικαστούν ασχέτως των σκεπτικών πεπιθήσεων. Οι χριστιανοί δελφοί στην Κένια ε, και η επίθεση εναντίον τους είναι ε, μια απόδειξη των εθνοτικών και θρησκευτικών ε, εντάσεων. Οι εθνοτικέ κοινότητες και οι ε, ένταση μεταξύ μουσουλμάνων και μη μουσουλμάνων στη χώρα είναι κάτι που το πετυχαίνουν οι τρομοκράτες με τη δράση τους διότι η κοινωνική περιθωριοποίηση, τα στερεότυπα, τα κοινωνικά όρια τους οδηγούν σε αυτή τη δράση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την κατάσταση διότι η καταπολέμηση του εκτρεμισμού δεν έχει να κάνει με τους μουσουλμάνους κατά των χριστιανών ή των ε, χριστιανών κατά των Εβραίων. Αφορά όλους τους πολίτες που δεν είναι εκτρεμιστές αλλά μετριοπαθείς. Πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις τάσεις και να σταθούμε ενωμένοι κατά του μίσους και της αδικίας. Πρέπει να δεχτούμε την πολυμορφία, να ενωθούμε και να προωθήσουμε τις αξίες της ισότητας, δημοκρατίας και ελευθερίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κλείνει η διαδικασία Κατστιάη. Να δώσω το λόγο στον κύριο Μίμητσα. Thank you, Madam President, members. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή αποδεικνύει παρόλο που υπάρχουν κάποιες κοινωνικές διαφορές, υπάρχουν κοινοί λόγοι που οδηγούν σε αυτή τη ριζοστικοποίηση. Η ανεργία, η φτώχεια, οι διακρίσεις, οι αποκλεισμοί θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ένα συντονισμένο και σοβαρό τρόπο η φτωχή, διεφθαρμένη, κακή διακυβέρνηση αποτελεί τον κοινό παρανομαστή. Οι κυβερνήσει πρέπει να αναλάβουν τι ευθύνε του. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη στηρίζει την χρηστή διακυβέρνηση, ε, δράσει που οδηγούν σε αυτήν και θα μπορούσαμε να κάνουμε και παραπάνω. Οι περιθωριοποιημένοι νέοι θα πρέπει να ξαναβρούν την αισιοδοξία τους και την αυτοεκτίμησή τους και όχι να θεωρούν πως έτσι χτίζουν τη φήμη τους και το όνομά τους. Θα πρέπει οι κυβερνήσεις να προσφέρουν την ε, εκπαίδευση και την παιδεία που θα οδηγήσει σε μια αξιοπρεπή ζωή και ε, στην εργασία. Η Γκαρίσα και τα γεγονότα εκεί αποδεικνύουν ε, για μια φορά ακόμα πως η παιδεία είναι η μεγαλύτερη απειλή για τους τρομοκράτες και για τη βία. Εμείς θα πρέπει να συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα, στο διεθνές επίπεδο, στο περιφερειακό αλλά και στο κοινοτικό επίπεδο για να αντιμετωπίζουμε τη ριζικοστικοποίηση των πληθυσμών και να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε κάποιες κοινέ δράσεις στα πλαίσια της στρατηγικής ασφάλειας έτσι ώστε να συντονιστούμε και να ολοκληρώσουμε τη μάχη κατά του βίου εξτρεμισμού και να θεωρήσουμε πως αυτό αποτελεί μια εγκάρσια προσπάθεια να γνωρίζω πως αντιμετωπίζουμε μια τεράστια πρόκληση και θα χρησιμοποιήσω κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας με τον πιο αποτελεσματικό και στοχευμένο τρόπο. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χθες για την οικοδόμηση δυναμικού για την ασφάλεια και την ανάπτυξη ενισχύει τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ ασφάλειας και ανάπτυξης. Οι ευρωπαϊκές αποκρίσεις θα συντονιστούν και θα έχουν πάντα μία διάσταση ασφάλειας και μία διάσταση αναπτυξιακή. Σε όλες τις ε, κρίσεις, τις σημερινές, τις μελλοντικέ και βεβαίως συμπεριλαμβάνεται αυτό και στη μάχη κατά της ε, εξτρεμιστικής βίας που ασκείται κατά των χριστιανών παγκοσμίως. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε 7 προτάσεις ψηφίσματος εδώ. Κλείνει η συζήτηση.